αυτή η οδηγία για την διασύνοριακή περίθαλψη. Ας μην ξεχνάμε το 40% του πληθυσμού βρίσκεται σε όμορες περιοχές και το ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι μόνο ένα 20% των πολιτών γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σε αυτό τον τομέα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να το προωθήσουμε. Επίσης χρειάζεται χρηματοδότηση του πακέτου αυτού για την υγεία. Κυρία Γκραπίνη, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Σας ευχαριστούμε. Τέλος, έχει μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας καθώς και τα εθνικά γραφεία πληροφόρησης. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα των ασθενών, ιδιαίτερα στις όμορες περιοχές. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη, διότι η ζωή και η υγεία είναι ύψης της σημασίας. Ευχαριστούμε. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπέλετ για την πολύ σημαντική έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαψη που τη θεωρώ πολύ σημαντική για μένα. Κάθε χρόνο εκατομμύρια Ευρωπαίων πηγαίνουν σε άλλες χώρες της Εύρωσης ε, με την επίγνωση και την βεβαιότητα ότι αν χρειαστεί μπορεί να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Ταυτόχρονα πολίτες ε, προγραμματίζουν να πάνε σε άλλα κράτη-μέλη. Γιατί, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δίνει την εγγύηση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη εκτός ε, της χώρας τους. Άρα είναι ασφαλέ να πούμε ότι η διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πολύ σημαντική για τους πολίτες της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεση και σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής διασυνοριακά. Πρέπει να τονίσω ότι συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Χρειάζεται δράση για τη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της οδηγίας. Και μάλιστα οι απόψεις είναι πολύ σημαντικές γιατί αντικατοπτρίζουν και την δική μας, ε, ε, τα δικά μας συμπεράσματα της Επιτροπής ε, σχετικά που δημοσιεύτηκαν το Σεπτέμβριο. Θέλω να, να ασχοληθώ εντάχει για το τι κάνουμε για να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Εμείς εξετάσαμε την ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες του ε, και λάβαμε δράση. Ξεκινήσαμε 26 διαδικασίες παραπομπής για καθυστερημένη ή ατελή ενσωμάτωση. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί τώρα και, μόνο οι, και όλες οι παραπομπές έχουν, στη φάση αυτή έχουν κλείσει. Η Επιτροπή προχώρησε σε, μια, ε, σε βάθος αξιολόγηση της συμμόρφωσης, εξετάζοντας προσεκτικά τα μέτρα που υιοθέτησαν τα κράτη-μέλη σε καθένα από αυτά. Η προσέγγιση αυτή δίνει αποτελέσματα. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη αλλάξει την εθνική τους νομοθεσία προς όφελος των ασθενών. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ωστόσο ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τον εντατικό διάλογο που έχει με τα κράτη-μέλη για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ενσωμάτωσης της οδηγίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οδηγία δίνει περιθώριο χειρισμών στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση. Ωστόσο, βλέπουμε στοιχεία διακρίσεων έναντι ε, πολιτών της Ένωσης που ζητούν θεραπεία σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, οι ασθενείς επίσης συχνά αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σύνθετες διαδικασίες εν ώψη θεραπείας στο εξωτερικό. Αναλαμβάνουμε δράση για να περιορίσουμε τις αδικαιολόγητες τέτοιες πρακτικές. Τον Ιανουάριο ξεκινήσαμε διαδικασίες παραπομπής κατά δύο κρατών μελών για τους εθνικούς κανόνες αποζημίωσης και επιπέδων αποζημίωσης. Επίσης καλωσορίζουμε την έκθεση για τα συστήματα αποζημιώσεων η έκθεση τονίζει την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών ε, όπως απαιτεί και η οδηγία. Η Επιτροπή θα συνεχίζει να ε, ενημερώνει τους πολίτες για τα δικαιώματά τους. Συμφωνούμε με τις συστάσεις της Επιτροπής σας επίσης ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για τα εθνικά, ε, για τα σημεία επαφής. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω κυρίες και κύριοι βουλευτές ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα εθνικά σημεία επαφής και θα δημιουργήσουμε και ένα scoreboard σχετικά για το στο εγγύς μέλλον. Η με τις προσπάθειες βελτίωσης αυτών των εθνικών σημείων επαφής τόσο ώστε να βελτιωθεί η ενημέρωση των ασθενών. Επίσης ενθαρρύνουμε τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών, μελών, κρατών μελών, ιδίω στις παραμεθόριες περιοχές. Και στο πλαίσιο αυτό εμείς υποστηρίζουμε τα ευρωπαϊκά δίκτυα τοπικών και περιφερειακών υγειονομικών αρχών για τη διαμόρφωση κοινών πλατφόρμων πολιτικής. Δύο σημαντικά σημεία θέλω να υπογραμμίσω στην έκθεσή σα. Την δημιουργία των 24 Ευρωπαϊκών Δικτύων αναφορά Ένα μείζον ζήτημα στην διασυνοδιακή συνεργασία, ιδίω για τι σπάνιε ασθένειε. Τα δίκτυα αυτά ωστόσο αντιμετωπίζουν προβλήματα, την ένταξή του κυρίω στα εθνικά συστήματα υγεία. Σα ευχαριστώ για την αίτηση, για το αίτημά σα, να υποστηρίξουν τα κρατημέλη το, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφορά ωστόσο. Δεύτερον, να συμφωνήσω ε, με την ε, πρότασή σας για τις ψηφιακές λύσεις. Εμείς υιοθετήσαμε μία σύσταση για το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Μητρό και, την, ε, το σχετικό έντυπο ανταλλαγή πληροφοριών, κάτι που επιτρέπει στα άτομα να έχουν πρόσβαση διασυνοριακά στα στοιχεία υγείας τους. Στην Εσθονία ξεκίνησαν πρόσφατα να, να ανταλλάσσουν και συνταγές με γειτονικά κράτη. Αυτό ενθαρρύνει και ενισχύει την προσβασιμότητα των ε, ιατρών και των ασθενών. Πιστεύω ότι η έκθεσή σας θα συμβάλλει σημαντικά στην σχετική συζήτηση. Προσβλέπω στην τελική σας έκθεση και σας διαβεβαιώνω ότι θα εξετάσουμε τις συστάσεις σας πολύ προσεκτικά. Η σύγκληση απόψεων μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων επιτρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά προ όφελο των ασθενών και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Και τώρα θα μιλήσουν πολιτικέ ομάδε. Το ΕΛΚ, ο κύριο Μπουσόη, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Ιβο Μπέλετ για την έκθεση. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που βοηθά τους ασθενείς για να τους να επιστρέφονται τα ιατρικά έξοδα σε άλλα κράτη-μέλη. Έχω υποβάλει τροπολογίες. Ε, ε, το 2010 2012 είχα υποστηρίξει αυτή την οδηγία και επίσης την είχα προωθήσει στη χώρα μου το 13-14. Ορισμένα κράτη-μέλη όμως έχουν ε, προβάλει διοικητικά μέτρα τα οποία αποτελούν πρόσκομα στην επιστροφή ιατρικών εξόδων. Επίσης, πολλοί ασθενείς δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους δυνάμει αυτής της οδηγίας. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Δυόμιση λεπτά ο κύριος Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς ε, να συγχαρώ τον κύριο Μπέλετ ε, και να τον ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε όσον αφορά τον στόχο αυτής της προσπάθειας. Θέλουμε να έχουμε την ευημερία των, ε, και το συμφέρον των ασθενών σε πρώτη γραμμή σε θέματα διασυνοριακά γιατί η διασυνοριακή παροχή υγείας δεν λειτουργεί απρόσκοπτα όπως θα έπρεπε. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να έχουν ε, πρόσβαση όλοι οι ασθενείς σε διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου και το κόστος της, ε, των διαφόρων θεραπείων να τους επιστρέφεται σε τελευταία ανάλυση. Δεν είναι δυνατόν να εξηγήσουμε ε, στους συμπολίτε μας ότι 26 από τα 28 κράτη-μέλη καθυστέρησαν τόσο πολύ όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας που ξεκίνησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαδικασίας παραβάση. Από το Ευρωπαρόμετρο ε, του 2015 φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας δεν γνώριζε καν Δύο χρόνια μετά την ε, εφαρμογή της ε, ε, οδηγίας, τα δικαιώματα που έχει. Η γνώση όμως αυτής της οδηγίας από τους συμπολίτε μας είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να εφαρμοστεί και στον τομέα της υγείας είναι περίπλοκη η πληροφόρηση και δεν είναι ικανοποιητική η πληροφόρηση που υπάρχει τώρα εδώ. Τα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν μέσω των εθνικών κέντρων επαφής. Αυτά τα κέντρα πρέπει να εξηγούν την κατάσταση σαφώς για όλους. Πρέπει να γίνει μια ευρεία εκστρατεία μέσω αυτών των ε, εθνικών σημείων επαφής για να γίνει γνωστή αυτή η οδηγία. Η σωστή πληροφόρηση είναι προϋπόθεση για να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό. Γι' αυτό απαιτούμε στην έκθεση και σωστά ακριβώς αυτό. Για την προστασία των καταναλωτών βεβαίως χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια και διαφάνεια και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξηγούν σαφώς τι υπηρεσίες προσφέρουν και σε τι περιπτώσεις και πώς επιστρέφονται τα έξοδα. Και η Κομισιόν ε, εξήγησε ότι η διαδικασία επιστροφής αυτών των εξόδων χρειάζεται ακόμη να βελτιωθεί πολύ. Από πλευρά της ομάδας μου τονίζω ότι πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση και για τις, ε, τους εμβολιασμού. Γιατί μειώνονται τα ποσοστά εμβολιασμών και αυτό δεν πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να το δεχόμεθα. Πρέπει να συμπληρωθεί η έκθεση στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρούπα, ECR. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας είναι μια μεγάλη ευκαιρία για πολλούς συμπολίτε μας που δεν έχουν την κατάλληλη ε, περίθαλψη στα κράτη τους. Η συνθήκη προβλέπει υψηλό επίπεδο ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όλων, αλλά η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα άτομα που ζουν σε μεθοριακές περιοχές, περιοχές στα παλιά κράτη-μέλη εποφελούνται από αυτή τη δυνατότητα. Κάποια άτομα επίσης πηγαίνουν σε φτωχότερες χώρες για να ε, τους ε, παρασχεθούν φτηνότερες υπηρεσίες υγείας. Πολλές χώρες υποφέρουν από το ότι οι πολίτες τους δεν έχουν πρόσβαση σε ε, ακριβές θεραπείες και φάρμακα. Χρειάζεται περισσότερη ευαισθητοποίηση φυσικά του κοινού. Αυτά τα εθνικά σημεία επαφή μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό όμω που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να βοηθήσουμε όσου υποφέρουν από σπάνιε ασθένειε να λαμβάνουν την κατάλληλη περίθαλψη. Και ναι, είναι επειδή είναι χαμηλός ο αριθμός ε, που πάσχει από κάθε μία από αυτές τις σπάνιες ασθένειες, ε, είναι δύσκολο να λάβουν τη σωστή περίθαλψη. Επίσης, πρέπει να γίνει έρευνα για νέα φάρμακα. Οι τιμές πολλών ε, από τα νέα φάρμακα, ωστόσο, είναι πολύ υψηλές. Αν υπάρξει μία πανδημία ή μία πολύ εκτεταμένη επιδημία, Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ο αναγκαίο εμβολιασμό για να αποφευχθεί αυτό, αλλά πρέπει να είναι ευθύνη των κρατών μελών αυτό. Ο κύριο Σελίμοβιτ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους Σκιώδης. Η ευρωπαϊκή διασυνοριακή περίθαλψη γίνεται το ένα και πιο σημαντική λόγω της μεγάλης κινητικότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλά γι' αυτό έχουμε και την υποχρέωση να βελτιώσουμε αυτό το πλαίσιο. Ένας βασικός τομέας είναι η διαφάνεια των φορέων παροχής υπηρεσιών, των φορέων υγείας. Θα πρέπει να ξέρω δηλαδή αν θα μου επιστραφούν τα έξοδα για να ξέρω κατά πόσο μπορώ να μεταβώ στο νοσοκομείο μιας άλλης χώρας. Επίσης υπάρχουν πολλές περιπλοκές στην επιστροφή εξόδων καθώς και ο μηχανισμός προσφυγών. Κανένας δεν θα επισκέπτεται νοσοκομεία σε άλλο κράτος μέλος εάν δεν ξέρει ότι θα του δοθούν σωστές απαντήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μια γενικότερη βελτίωση και ενόψη της παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κόνετσνα για ένα λεπτό από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο και τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τον συνάδελφο Μπέλε για τη θαυμάσια εκθεσή του, ιδιαίτερα για κάποιες ομάδες ε, ασθενών, αυτούς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες. Για αυτούς η κατάλληλη λύση είναι η διαμεθοριακή περίθαλψη. Πρέπει να υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι όμως και οι αναγκαίες γνώσεις, ιδιαίτερα για τις σπάνιες ασθένειες, γιατί αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, όπως είπα, εντός ενός κράτους μέλους. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες περίθαλψης που προσφέρει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των ειδών περίθαλψης που παρέχονται από τα διάφορα κράτη-μέλη και οι διοικητικές δυσχέρειες που δυσχεραίνουν την ε, εφαρμογή αυτή. Θα μπορούσε να βοηθήσει επίσης μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας. Αυτό που χαιρετίζω ιδιαίτερα είναι η έκκληση που γίνεται για να απλουστευθεί ε, η εφαρμογή της υποχρέωσης εμβολιασμού διότι σε ορισμένε ε, περιφέρειες διαπιστώνουμε ότι επανέρχονται ασθένειε που θεωρήσαμε ότι εδώ και πολύ καιρό έχουν εξαλειφθεί. Και πρέπει να ασχοληθούμε και με τις ε, αρνητικές, ε, τα αρνητικά εξατορικά στοιχεία της διαμεθοριακής συνεργασίας. Τι εννοώ, την παράλληλη επανεξαγωγή φαρμάκων το οποίο βεβαίως θίγει τα συστήματα υγείας των πιο φτωχών χωρών. Πρέπει να απογορευτεί αυτή η πρακτική. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πράσινου. Η κυρία Μέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ κύριε Μπέλετ για την εξαιρετική σας εργασία. Μόνο το 17% των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως προς την διασυνοριακή περίθαλψη. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί σε σχέση με τις παροχές στη διασυνοριακή περίθαλψη θα πρέπει να υπάρχουν σημεία διεπαφής των εθνικών αρχών. Όταν πρόκειται για την έρευνα, για παράδειγμα, ή την αντιμετώπιση των σπανίων ασθενειών. Γι' αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τα 30 εκατομμύρια πολιτών που πλήττονται από κάποια σπάνια ασθένεια. Βεβαίως χρειαζόμαστε δεδομένα, στοιχεία δηλαδή, για τις ασθένειες αυτές για να καταπολεμήσουμε και την απάτη. Αλλά ο ασθενής θα πρέπει να είναι στο κέντρο του γενικότερου μελήματός μας για να δούμε πώς μπορεί να ευεργετηθεί από αυτό το πλαίσιο. Νομίζω ότι όλοι έχουν δικαίωμα, ακόμα και αυτοί στους οποίους δεν, έχουν, δεν έχει χορηγηθεί άσυλο ή δεν έχουν χαρτιά. Η κυρία Μελέν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η διασυνοριακή κινητικότητα δίνει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες ε, οι οποίοι είναι δηλωμένοι και έχουν άδεια ε, διαμονής να μπορέσουν να μεταβούν αλλού. Και αυτό με σχετική ευκολία. Γι' αυτό και η οδηγία του 2011 για τη συνέχεια ιατρικής φροντίδας έχει μεγάλη σημασία. Πρόκειται για εθνική υπόθεση, αλλά θα πρέπει να αφορά όλα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να υπάρχει συμμεταχείριση σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα σύστημα υγείας παντού που ισχύει εδώ και 200 χρόνια. Θα πρέπει όμως να δούμε τι γίνεται ε, στην περίπτωση των μεταναστών και να έχουμε μία βάση δεδομένων ιδιαίτερα σε σχέση με τη χορήγηση αγχολητικών και τους εμβολιασμούς. Ο κύριος Πέτερλε για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Είναι ένα κείμενο που θα εξυπηρετήσει τους συμπολίτες μας. Είναι κάτι που το απαιτούν. Και για να μπορέσει επιτέλους να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, χρειάστηκε να εμπλακεί και το δικαστήριο για να μπορέσουν να ασκήσουν δηλαδή το δικαίωμά τους οι ασθενείς να θεραπευτούν σε μια άλλη χώρα και να τους επιστραφούν οι δαπάνες τους διότι πολλοί ασθενείς δεν υποφελούνται από αυτή την οδηγία και ε, εάν απευθυνθούν στον ασφαλιστικό τους οργανισμό έχουν δυσχέρειες για να τους επιστραφούν τα έξοδά τους αλλά δεν είναι τα μόνα προβλήματα αυτά δεν χρειαζόμαστε φυσικά μια νέα οδηγία. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε να εφαρμοστεί υπάρχουσα. Η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγεία θα <coughs> καταστεί δυνατή μόνο τότε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάλη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα από τα βασικά πλονεκτήματα της Ενωμένης Ευρώπης είναι το δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη κάθε κράτους μέλους. Το δικαίωμα, ιδίως δεν το δικαίωμα αποζημίωσης για τυχόν θεραπεία εκτός του κράτους μέλους. Αυτό γίνεται σημαντικότερο τώρα που ζούμε σε μία περίοδο γρήγορης εξέλιξης ασθενειών. Είναι ευθύνη μας λοιπόν να παρέχουμε ίση πρόσβαση σε όλα τα υγειονομικά συστήματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Για να γίνει κάτι τέτοιο, ωστόσο, πρέπει να υπάρχει το σωστό πλαίσιο. Να διευκολύνουμε την αυξημένη συνεργασία σε διάφορους τομείς της ιατρικής και υγειονομικής περίθαψης. Για παράδειγμα, θέλω να αναφερθώ στο e-health ή την θεραπεία σπάνιων νόσων. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο ασθενείς, αφορά όλους. Μιλάμε κατά συνέπεια για την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι πόσοι πολίτες ξέρουν τα δικαιώματα αυτά. Ιδίω δε το δικαίωμα να λάβουν αποζημίωση αν τύχουν ε, περίθαλψης εκτός κράτους μέλους. Μια τελευταία παρατήρηση. Αυτό το τελευταίο δείχνει την ανάγκη να μπορούν τα κράτη-μέλη να ενημερώσουν σωστά τους πολίτες για τα δικαιώματά τους. Κύριος Μαριάς. Η διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οπωσδήποτε συνιστά ένα από τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παλαιότερα είχαμε την ε, δυνατότητα και την προσπάθεια θα έλεγα διαφόρων ασθενών να πάνε σε άλλο κράτος της ευρωπαϊκής ένωσης όπου εκεί γινόταν ε, επεμβάσεις ε, και όπου στη χώρα τους δεν μπορούσε να παρασχεθεί συγκεκριμένη περίθαλψη. και αυτή ήταν η γενική τάση αλλά βεβαίως υπήρχε τεράστιο πρόβλημα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα έπαιρναν οι ασθενείς τα ποσά τα οποία είχαν πληρώσει τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει και οι ασθενείς πηγαίνουν σε χώρες όπου είναι πιο φθηνή η ίδια η περίθαλψη. νομίζω ότι η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί. αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε επίτροπε κύριε Ανδρουικάιτης για το θέμα της επιδημίας της γρίπης στην ελλάδα έχουμε πάνω από 39 νεκρούς. Υπάρχει μια τεράστια επιδημία γρήπης και θα ήθελα να ρωτήσω εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σας έχει ζητήσει τη βοήθεια και τι θα γίνει με την έλλειψη εμβολίων που υπάρχει για την αντιμετώπιση της γρήπης. Θέλουμε μια απάντηση στο θέμα αυτό γιατί απασχολεί τον ελληνικό πληθυσμό. Ευχαριστώ. Κύριε Πέτικα, ένα λεπτό. Η διασυνοριακή περίθαλψη είναι σημαντική και θα γίνεται όλο και σημαντικότερο, και σημαντικότερο στο μέλλον. Και από την οπτική της υγείας των πολιτών και από την οπτική της μείωσης των πόρων. Η περίθαλψη πρέπει να προσφέρεται σε ασθενείς που το χρειάζονται και που και πρέπει να υπάρχουν και επαρκή πόροι σε εθνικό επίπεδο για την κάλυψη αυτών των δαπανών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέλετ, τον εισηγητή, και την Επιτροπή που ήταν εξαιρετικά δραστήρια στο σημείο αυτό. Είναι κρίμα το ότι τόσα κράτη-μέλη δεν έχουν ενσωματώσει την οδηγία σωστά στο εθνικό τους δίκαιο. Ιδίως δεν έχουν ενημερώσει τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, ενώ δεν αποζημιώνουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρόκειται για ένα πολιτικό παιχνίδι στις πλάτες της υγείας των πολιτών. Πρέπει να αναλάβουμε δράση στο σημείο αυτό το συντομότερο δυνατό, φέρνοντα τα κράτη-μέλη ενώπιον τη δικαιοσύνη, αν χρειαστεί. Κύριε Καπεθόνου ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διασυνοριακή υγεία είναι ελεύθερη κυκλοφορία. Το Ευρωβαρόμετρο θέτει την υγεία ως ένα από τους βασικούς, ε, ε, μία από τις βασικές αξίες της, ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλά η εθνική υγεία είναι εξαιρετικά εθνικοποιημένη ακόμα. Η οδηγία είναι μια εξαιρετικά φιλόδοξη. Η εφαρμογή της ωστόσο ήταν άνηση από κράτη-μέλη. Ξεκινώ προσθέτοντας ότι για την επιτυχία της οδηγίας αυτής χρειάζεται μία βάση, μία δέσμευση των κρατών μελών με τα εθνικά υπέρ του εθνικού συστήματος υγείας και υπέρ της ενίσχυσής τους. Αυτό μπορεί να ενσωματώσει, δεν μπορεί να αλλάξει και πρέπει να ενσωματώνει και τη διασυνοριακή διάσταση. Θα σας παρακαλούσα να μιλάτε λίγο πιο αργά. Προχωρώ. Ε, λέω ότι αυτό θα πρέπει να προχωρά βήμα-βήμα, στόχο-στόχο. Με την ευρωπαϊκή ταυτότητα υγείας. Με την αποφυγή των διακρίσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο και με την εφαρμογή της καθολικότητας της υγείας επιτρέποντας σε όλους τους πολίτες να έχουν την καλύτερη δυνατή υγεία. Δεύτερον, αναγνώριση της συνταγής. Τρίτον, η οδηγία θα πρέπει, και πρέπει να προχωρήσει και ένας νέος στόχος της Επιτροπής είναι η ψηφιακή υγεία. Τα δημόσια συστήματα υγείας είναι οι μόνοι που εξασφαλίζουν τα στοιχεία της ιδιωτικότητας και της δικαιοσύνης του συστήματος υγείας. Σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα λοιπόν που ξεκινάει η Επιτροπή ζητώ να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στους δημόσιους οργανισμούς των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Γκέρικε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόεδρε, η έκθεση ε, εφαρμοστικών διατάξεων δείχνει ότι μπορούμε να ελέγξουμε την νομιμότητα του πλαισίου φαρμακο, θρησκευτικής ε, διασυνοριακής περίθαλψης. Αυτό αφορά και ιδιαίτερα τις σπάνιες ασθένειες. Γι' αυτό οι πολίτες θα πρέπει να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματα τους ε, δυνάμει της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει μία εκστρατεία πληροφόρηση σε σχέση και με τα εθνικά σημεία επαφής με συναφείς πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει ένα γενικό πλαίσιο πληροφοριών στα εθνικά σημεία επαφής για τους πολίτες που θέλουν να λάβουν διασυνοριακή περίθαλψη. Λίζε για ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι κύριε Επίτροπε, όταν ε, είναι κανείς, ε, έχει κανείς γενέθλια ή την πρωτοχρονιά, τι τους ευχόμαστε στους ανθρώπους. Υγεία. Η υγεία λοιπόν πρέπει να είναι πιο πολύ στο κέντρο της πολιτικής και της Ένωσης. Στο βαθμό της ε, αρμοδιότητάς μας. Αλλά υπάρχουν αρκετά σημεία για τα οποία έχουμε αρμοδιότητα. Για το ΕΛΚΑ είναι κεντρικό θέμα αυτό. Πρόσφατα, με πρόταση του Προέδρου μας, Μάνφρετ Βέμπερ, εκπονήσαμε ένα κείμενο για την καταπολέμηση του καρκίνου, έχει και πολύ προσωπικά αίτια πίσω. Στο έγγραφο αυτό γράφουμε από τη μία ότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε με βάση αρμοδιότητές μας, το ώστε σε 20 χρόνια να μην πεθαίνει κανείς από αυτή την ε, φοβερή ασθένεια και ε, αναφέραμε πολλά σημεία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα ορίζον Ευρώπη ο καρκίνος και ιδιαίτερα ο παιδικός καρκίνος πρέπει να αντιμετωπιστεί περισσότερο και λέμε ακόμη ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών να εφαρμοστεί καλύτερα. Γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Ιβο Μπέλετ που ε, εκπώνησε αυτή την έκθεση και ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια με ευρία πλειοψηφία, με ευρύτατη πλειοψηφία. Τα κράτη-μέλη πρέπει να σταματήσουν να σκέφτονται μόνο το βραχυπρόθεσμο κόστος. Ο ασθενής πρέπει να είναι στο κέντρο της εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Η έκθεση είναι η σωστή έκκληση προς τα κράτη-μέλη να σκεφτούν τα συμφέροντα του ασθενούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Να περάσουμε τώρα στο Catch Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Φαγία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιβο Μπέλετ καταρχήν. Η, ε, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα πρέπει να διέπεται από αλληλεγγύη. Γι' αυτό η οδηγία αυτή δίνει πολλές ελπίδες, αλλά δυστυχώς οι ασθενείς δεν ξέρουν καν για την ύπαρξή της και οι επαγγελματίες δεν την χρησιμοποιούν. Επίσης υπάρχουν ε, προσκόμματα στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Δεν μπορούμε όμως να την πετάξουμε στο κάλαθο των χρήστων γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να λειτουργήσει αυτή η οδηγία ιδιαίτερα για τους ασθενείς που έχουν σπάνιες ασθένειες, ιδιαίτερα ογκολογικής φύσης. Θα πρέπει να υπάρχει γνώση για την ύπαρξη αυτής της οδηγίας, καθώς και να γνωρίζουμε ποια είναι τα κέντρα εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλεκτρονική υγεία επίσης θα βοηθούσε ιδιαίτερα, αλλά η ηλεκτρονική υγεία θα πρέπει να είναι ενιαία και να αφορά προγράμματα ιδιαίτερα στον, ως προς τον εμβολιασμό. Κύριε Φαρία, μιλήσατε πολύ γρήγορα. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολο το έργο των ε, διερμηνέων. Κύριος Ρέντμαν. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω το γεγονός ότι ε, λαμβάνουμε γνώση τα πλαίσια λειτουργίας της διασυνοριακής περίθαλψης. Συμφωνώ με τον εισήγητη, αλλά εδώ και οκτώ χρόνια έχουμε εγκρίνει την οδηγία και οι πολίτες δεν ξέρουν ότι μπορεί να έχουν επιστροφή ιατρικών εξόδων ακόμα και αν η περίθαλψη έγινε σε ένα άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει να γίνουν ειδικέ εκστρατείες για την ύπαρξη εθνικών σημείων επαφής και ανταλλαγής πληροφοριών. Υπάρχουν ε, πολλά διοικητικά προσκόμματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, διότι όλα σχετίζονται με την ε, ε, λανθασμένη μεταφορά της οδηγίας. Η επιστροφή εξόδων θα πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία fast check. κυρία Βάουτμαντς, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε ένα σημαντικό θέμα διασυνοριακές ε, υπηρεσίες υγείας. Και συγχαίρω τον συνάδελφό μου από την περιοχή του Λιμβούργου, τον Ιβο Μπέλετ, για αυτή τη θαυμάσια έκθεση. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ουσιώδε το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι πολλοί συμπολίτε μα δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά του, όπω δείχνει και το Ευρωπαρόμετρο. Το 2015 μόνο 20% των συμπολιτών μα γνώριζαν το δικαίωμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενημερώσουμε του πολίτε για τα δικαιώματα αυτά που έχουν. Ο στόχος είναι να τους παράσχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες υγείας. Όταν είναι κανείς άρρωστος, θέλει να γίνει καλά. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες. Θεωρώ ότι το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η γραφειοκρατία ε, δυσχεραίνει την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις συστάσεις να υπάρχει μόνο μία θηρίδα όπου να απευθύνονται οι πολίτες που να τους παρέχει όλες τις σωστές ταχείες προφορίες. Ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ, Madame la ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υγεία αποτελεί για τον άνθρωπο το πολυτιμότερο αγαθό και πρέπει να προστατεύεται με κάθε τρόπο. Παράλληλα, η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης ε, παρέχει τη δυνατότητα σε πολλούς ασθενείς να ε, εξασφαλίσουν η υγειονομική περίθαλψη όχι μόνο στη χώρα τους αλλά και σε άλλα κράτη μέλη της ε, ευρωπαϊκής Ενώσης κυρίως τα όμορα. πρέπει λοιπόν τα κράτη να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να διευκολύνουν την ε, ομαλή ε, κινητικότητα των ασθενών προς άλλα κράτη. προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει η αντιμετώπιση διαφόρων γραφειοκρατικών μεθόδων απλοποίηση ορισμένων διοικητικών μέτρων καθορισμός των αποζημιώσεων καθώς επίσης και προσπάθεια για την αντιμετώπιση της απάτης των επιδημιών και κυρίως της ε, ε, υγειονομικής περιθάλψης των παρανόμων μεταναστών οι οποίοι πολλές φορές συσσωρεύονται όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ελλάδος σε μεγάλους αριθμούς ε, στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες. Ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ζω στην σε μεθοριακή ζώνη που συνορεύει με το Βέλγιο και πολλοί άνθρωποι από το Βέλγιο πολύ απλά πάνε στον γιατρό στη Γερμανία. Έτσι ήταν τα πράγματα, αλλά πλέον δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια συμφωνία στις μεθοριακές περιοχές που λέγεται Ίζομ και με αυτήν μπορούσε να πάει χωρίς διατυπώσεις ο Βέλγος στο Γερμανό γιατρό. Ε, τώρα το κατέργησαν αυτό και βεβαίως να πούμε εδώ πέρα ότι είναι ελαφρώς αδιάφορο το ποιες ε, είναι οι διατυπώσεις μεταξύ των ε, ταμείων. Θέλει τον καλύτερο γιατρό ή δυνατόν στη γλώσσα του. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Και βεβαίως ε, λέμε πάρα πολύ συχνά το τι γίνεται, αλλά έχουμε εδώ πέρα ένα θαυμάσιο παράδειγμα στις μεθοριακές αυτές τις περιοχές και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το προωθήσετε και αν δεν ε, γίνεται να το κάνετε υποχρεωτικό. Αν οργανωθούμε έτσι νομίζω θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Σας ευχαριστώ. Λένε βεβαίως ότι πρώτα η υγεία και έχουν ε, δίκιο και ειδικά στην ε, σύγχρονη κοινωνία με την οικονομία μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουν οι πολίτες πρόσβαση στην υγεία όσο το δυνατόν πιο εύκολα γιατί είναι άλλο βεβαίω να έχει κανεί πρόσβαση όταν είναι υγιής, αλλά όταν είναι άρρωστο, οποιαδήποτε επιπλέον γραφειοκρατία κάνει τα πράγματα δύσκολα. Γι' αυτό ακριβώ ε, η οδηγία αυτή είναι τόσο σημαντική. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει περισσότερες πληροφορίες, ειδικά σχέση με διάφορες εκστρατείες για την μείωση της ε, γραφειοκρατίας. Γιατί υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει βοήθεια, αλλά συχνά είναι δύσκολη η πρόσβαση. Αυτό πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος. Ο κύριος Λίζε μίλησε για την καταπολέμηση του καρκίνου εγώ στο μεσημεριανό διάλειμμα θα πάω σε μια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Επιληψία. Πολλά συμβαίνουν λοιπόν και πρέπει να τα μάθουν οι πολίτες. Και τέλος ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο, τον κύριο Ιβο Μπέλετ, τον εισηγητή. Ε, μπορείτε να του το πείτε βεβαίω, Σας ε, ευχαριστώ κύριε Αντριοκάητης, μπορείτε να ολοκληρώσετε την συζήτηση πριν από τον κύριο Μπέλετ βεβαίω. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που σας άκουσα και σας ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Να επαναλάβω και πάλι ότι τώρα είναι μια καλή στιγμή για όλους μας να ενημερώσουμε τον κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινήσει αυτή η εκστρατεία, γιατί έρχονται και ευρωεκλογές πρέπει να παραμείνουν αυτά τα ζητήματα ψηλά στην ατζέντα και σας παρακαλώ όσοι τώρα θα βγείτε για προεκλογική εκστρατεία και θα παρουσιάσετε τα προγράμματα στον κόσμο να τα λέτε αυτά. Βεβαίως βλέπω κάποιες αντιπαραθέσεις ε, ε, όσον αφορά την ε, επικουρικότητα μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί υπάρχει τόσο χαμηλή ενημέρωση. Μα αν ρωτήσετε τα κράτη-μέλη θα σας πούνε ναι, είναι εθνική αρμοδιότητα και υπάρχει αυτή η εποδός. Αν δείτε λοιπόν την αξιολόγηση που υπάρχει θα δείτε ότι δεν θέλουν να κάνουν περισσότερα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών. Γιατί, Γιατί υπάρχει μια λάθος αντίληψη για την επικουρικότητα. Αν λοιπόν ε, κάποιοι ε, μπορούν ε, να αντιμετωπιστούν σε κάποια άλλη χώρα. Ας γίνει αυτό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει και η νοοτροπία. Δεν, ανάγκη να, δεν χρειάζεται μόνο να έχουμε κάποια υποδείγματα και να έχουμε εκεί πέρα στα έγγραφα τα σημεία επαφής. Πρέπει να αλλάξει το όλο αφήγημα και η σκέψη των ε, κυβερνήσεων. Λοιπόν, η σύγκληση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς ε, προσπαθούμε ακριβώς να καταργήσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν στον τομέα της υγείας και υπάρχουν κάποιοι βασικοί πυλώνες ε, στον τομέα των χρεώσεων, των επιστροφών, ε, την πρόσβαση στα διοικητικά δεδομένα, τις ε, διοικητικές διαδικασίες και άλλα τέτοια ζητήματα. Σας διαβεβαιώ πως η Κομισιόν θα εξετάσει το πώς ακριβώς θα προωθήσει αυτήν την έκθεση όταν εγκριθεί. Θα αναλάβουμε δράση αν ε, δεν τηρηθεί το πνεύμα και το γράμμα εδώ της ε, νομοθεσίας και ακριβώ ε, θέλουμε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των ασθενών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για τη δουλειά που έχει κάνει στο θέμα. Συγκεκριμένα θα ήθελα να εξάρω την αναφορά της Προέδρου της Αρμόδιας Επιτροπής, του Αντιπροέδρου του κυρίου Γιάβορ, και του κυρίου Μπέλετ και των σκιωδών εισηγητών. Κάτι λοιπόν το οποίο μπορεί να έχει ένα πρακτικό αντίκτυπο ε, είναι αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, και κάτι άλλο. Ε, επειδή υπήρχε ένα ερώτημα από τον κύριο Μαριά για την γρήπη στην Ελλάδα. Μα σε όλες τις χώρες είναι αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πως έχουμε αρκετά εμβόλια για την εποχιακή γρήπη, αλλά η επιδημία της γρήπης υπάρχει γιατί ο κόσμος δεν εμβολιάζεται το εμβόλιο, υπάρχει και στην Ελλάδα. Επαφείτε τώρα σε ελληνικές αρχές να κάνουν περισσότερα και να ενημερώσουν τον κόσμο. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που είναι κατά των εμβολίων με την θανατηφόρα εκστρατεία τους. Σας παρακαλώ λοιπόν εμβολιαστείτε και κάντε και εκστρατεία υπέρ των εμβολίων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλετ θα κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά την τελευταία παρατήρηση του κ. Μαριά, να προσθέσω ότι υπάρχουν προτάσεις, ε, υπήρχαν προτάσεις ε, να συμπεριληφθεί ε, και, η, και ο εμβολιασμό σε αυτήν την οδηγία, αλλά η ομάδα του κ. Μαριά, η ΕΣΥΑ, είχε διαφωνήσει. Ε, Τέλο πάντων, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ όλους σας. Ε, ευρία στήριξη αυτού του κειμένου Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτρόπε που αναφερθήκατε στο γεγονό ότι θα εντείνετε τις προσπάθειές σας για την απλοποίηση των διαδικασιών αφενός και αφετέρου ότι σκοπεύετε να ενισχύσετε τα σημεία επαφής. Σημαντικός ο ρόλος τους, θα στηρίξουμε την προσπάθειά σας. Και ελπίζω να ακούσουν όλοι το μήνυμά σας. Ρόλος των Ευρωβουλευτών είναι αυτό το μήνυμα να το προωθήσουν και να το προβάλλουν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και αργότερα. Δεν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα απαραίτητα στους ασθενείς να παίρνουν τα σύνορα, αλλά ειδικά για ασθενείς ε, με χρόνια νοσήματα, με σπάνια νοσήματα και για ασθενείς σε μεθοριακές περιοχές ε, είναι χρήσιμη αυτή η δυνατότητα και ενδεχομένως και πιο οικονομική. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη εξυπηρετεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών. Το είπε και ο Πίτερ Λίζε και άλλοι. Αυτό δεν κοστίζει χρήματα. Το θέμα είναι να γίνει σωστή εφαρμογή αυτού του, οργάνου, αυτού του εργαλείου, αυτής της οδηγίας, για να δείξουμε την πρόσθετη αξία, την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Τελειώνοντας, να πω κυρία Πρόεδρε, ότι θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στη Μαρία Γκραπίνη που είναι συνεισηγήτρια από την Επιτροπή ΕΜΚΟ και ε, τις ευχαριστίες μου στους κοιόδης συγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έκλεισε αυτή η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει ευθύ αμέσω. Να ξεκινήσουμε, αφήνουμε τους επιτροπούς να πάρουν θέση. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση τη κυρία Μποναφέ για τι ελάχιστε απαιτήσει για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Κυρία Μποναφέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω τους και όλους για τη συνεισφορά τους στην τόσο σημαντική συζήτηση τους τελευταίους μήνε εργασία μα. Θα ξεκινήσω από ένα δεδομένο. Μόνο το 2017 οι συλλογικές ε, λογές νερού ήταν περίπου 6 ε, κυβικά χιλιόμετρα. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να διπλασιαστεί ως το τέλος της χρονιάς. Εδώ υπάρχει θέμα διεθνούς ανταγωνισμού για την ε, υδροδότηση, την παροχή του νερού και τη χρήση των υδάτινων πόρων. Αυτό έχει επιπτώσει στην οικονομία, στη ζωή των κοινοτήτων και στα οικοσυστήματα από τα οποία εξαρτώνται οι ίδιες οι κοινότητες, οι πολίτες. Και βεβαίως αυξάνεται η ζήτηση. Οι επιπτώσει των κλιματικών αλλαγών γίνονται όλο ένα και πιο προφανεί. Αυτό μα φέρνει αντιμέτωπου με την πιθανότητα οι περιοχέ που έχουν προβλήματα λειψιδρίας ή ξηρασία να είναι περισσότερε στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε την όλο ένα και πιο πιεστική ανάγκη ορθή και αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων, του νερού, που θεωρείται ένα πολύτιμο αλλά σπάνιο αγαθό. Α είμαστε σαφεί. Η Ευρώπη δεν είναι, δεν είναι μια ήπειρο ε, χωρί νερό. Όμως ε, ε, η δροδότησή μας μας ανησυχεί και είναι ανησυχητική τουλάχιστον για το μισό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ να σας δώσω πάλι κάποια δεδομένα. Η έλλειψη νερού, η λειψιδρία, είναι ένα θέμα που αφορά ήδη το 11% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 17% της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Φύρου. Από το 1980 ο αριθμός περιπτώσεων λειψιδρίας στην Ευρώπη αυξήθηκαν και έχουν επιδεινωθεί οι σχετικέ ε, καταστάσει. Το κόστο υπολογίζεται σε 100 δι ευρώ τα τελευταία 30 χρόνια. Η μόνη λειψιδρία του μόνο, μόνο, 2017 έδειξε πόσο σημαντικέ είναι οι οικονομικέ απώλειες αυτού του φαινομένου. Αυτό το δείχνει και η μελέτη εντεκτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά για τον τομέα τη γεωργία στην Ιταλία, α πούμε, όπου υπολογίστηκαν 5 δις ευρώ οι απώλειες. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η έλλειψη νερού, η λειψιδρία, δεν περιορίζεται μόνο σε, μια πολύ συγκεκριμένη, σε πολύ συγκεκριμένο αριθμό περιοχών τη Υπήρου που βρίσκονται όλε στο νότο τη Ευρώπη. σα ίσα αφορά ολόκληρο το χώρο, την επιφάνεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δική μα ευθύνη λοιπόν είναι να βρούμε κατάλληλε απαντήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διατηρήσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό για του πολίτε και να προφυλάξουμε και το περιβάλλον. Το σημείο θετηρία θα πρέπει να είναι αυτό του η αρχή τη κυκλική οικονομία να ισχύσει και εδώ. Ένα νέο μοντέλο μοντέλο ανάπτυξη στην Ευρώπη ε, και να ισχύσει και για του υδάτινου πόρου να υπάρχει εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση μέσω ενό νομοθετικού εργαλείου που να είναι συγκεκριμένο προ αυτό το σκοπό. Για να ε, εγγυηθεί την νομοθετική σταθερότητα που θα ευνοήσει τι επενδύσει σε αυτό τον τομέα που είναι πολύ σημαντικέ. Σημαντικέ για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα. Υπάρχει ήδη μια οδηγία πλαίσιο για το νερό, για του υδάτινου πόρου, που αναφέρει την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων ω ε, συμπληρωματικό μέτρο για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των υδάτινων πόρων. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφέ. Λείπει συγκεκριμένη νομοθεσία με ξεκάθαρους κανόνες ώστε να μπορούμε να υποφεληθούμε πλήρως από τις ε, δυνατότητες αυτού του εργαλείου βάσει των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δυναμικό της επαναχρησιμοποίησης του νερού μέχρι το 2025 είναι 6,6 ε, δις ε, κυβικά μέτρα σε σύγκριση με το τωρινό 1,1 κυβικών μέτρων νερού το χρόνο, 1,1 δις. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Γι' αυτό η, Ευρωπαϊκή, Επιτροπή ΕΝΒΗ υποστήριξε με μεγάλη πλειοψηφία τον κανονισμό όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, τον ένταξε στο ε, πλαίσιο τη όλη αλλαγή που θα φέρει η κυκλική οικονομία. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να, πετύχει, να επιδιώξει του στόχου τη κυκλική οικονομία με τον ορισμό, με εναρμονισμένων μέτρων σε επίπεδο ευρωπαϊκό για να διασφαλίσουμε την επιστη, μα ε, επάρκεια στο εσωτερικό της Ένωσης. Ως Επιτροπή ΕΝΒΗ συμμεριζόμαστε το γενικό σχέδιο και την γενική πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι ακριβώς αξιοποιεί τις εμπειρίες της, ε, των εθνικών νομοθεσιών, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και τα πειράματα που έγιναν εκεί. Θα πρέπει λοιπόν ως Κοινοβούλιο να συμμετάσχουμε με κάποιες τροπολογίες ώστε να είναι αποτελεσματικότερη νομοθεσία κατά την απόψή μας, ιδίως προς τους ορισμούς, τους ρόλους και την αρμοδιότητα των διάφορων φορέων που θα εμπλέκονται εδώ, καθώς και τι βασικέ δραστηριότητες διαχείριση του κινδύνου. Εντάχει, περισσότερε λεπτομέρειε, Θεωρήσαμε σημαντικό να οριστεί καλύτερα ε, το ποιοι είναι οι βασικοί φορείς που θα ασχολούνται με την ε, επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων και πώς θα δημιουργηθούν οι εγκαταστάσει επεξεργασίας, που θα είναι ο τελικός χρήστης και ταυτόχρονα διαχειριστής του δικτύου, ε, των δικτύων αγωγών και αυτό που θα ασχολείται με τη συλλογή των νερών, προ των υδάτων και λιμάτων προ επαναχρησιμοποίηση. Βάσει των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει τη μελέτη του GRC, θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε και με τον παράμετρο τη Αλμονέλα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη επιστημιστική ασφάλεια για του πολίτε. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίση να δοθεί στην ανάγκη ε, μέτρων ευαισθητοποίηση που θα φωτίζουν κυρίω το πόσο σημαντικό είναι να εξοικονομείται ε, το νερό στη χρήση του και ότι η επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων δεν θα φέρει επιπτώσει στην υγεία των ανθρώπων και ζώων. Το Κοινοβούλιο κλείνει τώρα τη διαδικασία τη πρώτη ανάγνωση. Είμαι βέβαια ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να βρει μια κοινή θέση που θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να ξεκινήσει αμέσω τη διαδικασία των τριμερών διαλόγων για να εγκριθεί αυτή τόσο σημαντική νομοθετική πράξη. Ευχαριστούμε κυρία Βέλα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω, τη Σιμώνα Μποναφέ για την ε, πολύ καλή δουλειά που έκανε όπως και οι σιχειώδεις ηγητές για αυτή την οδηγία. το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι κρίσιμο προκειμένου να προχωρήσει το θέμα αυτό στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Όπως είπε η Σιμώνα, το είδωρ είναι πολύτιμο ε, Πολύτιμο πόρος και χρησιμοποιείται και τόσο από την κατανάλωση από τους ανθρώπους και στη βιομηχανία, στη γεωργία κλπ. Παρ' όλα αυτά γίνεται όλο και πιο σπάνιος πόρος. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε προβλήματα έλψης όλο το χρόνο. Το 2018 το καλοκαίρι καταλάβαμε ότι το νερό γίνεται ανησυχία για πολλά κράτη-μέλη, ακόμα και για αυτά που συνήθως δεν συνδέονται με λειψιδρία ή ξηρασία. Αυτά τα προβλήματα πιθανότατα θα χειροτερεύσουν κυρίως εξαιτία της κλιματική αλλαγής. Μαζί με τα μέτρα αποδοτικότητα στη χρήση του νερού, ε, η μείωση της κατανάλωσης, η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να αποτέλεσε και αυτή μια λύση, καθώς επίσης και μια ε, ολοκληρωμένη πολιτική χρήση των υδάτων. Ε, το συγκεκριμένο κείμενο προτείνει την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ως αξιόπιστη ε, πολιτική, αξιόπιστη μέθοδο εξοικονόμησης υδατός στην γεωργία κυρίως. Αυτό έρχεται να δέσει με την κυκλική οικονομία την οποία προωθούμε τόσο πολύ. Ο στόχο είναι να διευκολύνουμε την αναχρησιμοποίηση νερού στη γεωργία όπου αυτό είναι ασφαλές, ε, ε, δυνατό και οικονομικά αποδοτικό. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τα συμφέροντα του καταναλωτή και τα συμφέροντα του περιβάλλοντος ταυτόχρονα. Οι εναρμονισμένες ελάχιστες παράμετροι θα βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα και θα δημιουργήσουν και καινούργιες εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσήλωσή του και για την πρόοδο που έκανε μέσω αυτής της έκθεσης. Αναμένουμε έναν καρποφόρο διάλογο. Ευχαριστώ. Κυρία ένα λεπτό εκ μέρους Επιτροπής Άγκρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τώρα κλείνει το κενό αυτής ε, της ε, νομοθεσίας όσον αφορά την πίεση που υφίστανται η ΙΔΑ, την υπόρρη λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Γι' αυτό έχει σημασία ακριβώς ο βιολογικός καθαρισμός και η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Έχουμε λοιπόν μία επέκταση του πεδίου εφαρμογή από την οδηγία και σε άλλους τομείς. Έτσι σας υπενθυμίζω ότι η Γεωργία έχει ήδη πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές, παραδείγματος χάρη τον κανονισμό περί τροφίμων που αναφέρει ξεκάθαρα το τι πρέπει να γίνει με τα χρησιμοποιημένα υδατά και έχει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για να είναι ασφαλή και τα γεωργικά προϊόντα. Η εφαρμογή αυτού του κανονισμού σημαίνει πολλά πλέον αλλά δεν θα πρέπει να επιβαρύνει περαιτέρω τους αγρότες. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις των ομάδων. Για το ΕΛΚΑ, για ένα ο κύριος Καμπούς. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μποναφέ για το έργο της και για την ε, καλή συνεργασία με τους ε, σκιώδες ηγητές. Ο κανονισμός το οποίο θα ψηφίσουμε σήμερα θα βοηθήσει και στην ε, καλή χρήση του υδατός, τη βιώσιμη χρήση του υδατός, αλλά και στην πρόθεση της κυκλικής οικονομίας. Θα πρέπει να έχουμε... Συζητώ συγγνώμη από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε μετάφραση στα αγγλικά, διακόπτη πρόεδρος. Ωραία, μπορείτε να συνεχίσετε. Παρόλο ότι ο κανονισμό περιορίζεται στι γεωργικέ χρήσει του νερού, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ξεκαθαρό ότι η διεύρυνση αυτή τη μεθόδου θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού ε, και για άλλου τομεί. Η συγχρηματοδότηση μέσω ενό προγράμματο LIFE για προγράμματα αναχρησιμοποίησης του ύδατο σε βιομηχανικό ε, περιβάλλον της Ταραγώνα είναι πάρα πολύ σημαντικό για παράδειγμα ε, ω πρόγραμμα πιλότο. Από ό,τι φαίνεται το 2030 ο, το, το 50% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάσει από λειψιδρία. Σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτό μπορεί να μην φαίνεται πρόβλημα, αλλά Κάνω έκλειστο στο Συμβούλιο για να καταλάβει ότι αυτό που επηρεάζει σήμερα τις χώρες του Νότου της Ευρώπης αύριο θα επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Οπότε στο μέλλον είναι σημαντικό η Κομισιόν να προτείνει αυτό που είναι κανονισμός σήμερα να γίνει με ε, οδηγία στο μέλλον έτσι ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε προκαταβολικά και όχι εκ των υστέρων. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για ένα λεπτό η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ θερμά την συγγήτρια την κυρία Μποναφέ. Είναι ειδική σε αυτό το θέμα και για την ε, κυκλική οικονομία και είναι πολύ σημαντικό που το θέμα της επαναχρησιμοποίησης των ε, υδάτων μπαίνει μέσα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Συγχαρητήρια κυρία Μποναφέ. Στην Ισπανία Είμαστε, η Ισπανία μάλλον είναι η χώρα η οποία πιο πολύ επαναχρησιμοποιεί τα ύδατά τη. Αυτό για ιστορικού λόγου. Όμω αυτό είναι και πάλι πολύ ευαίσθητο. Ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ασταθή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η, ο υδροφόρο ορίζοντα στην Ισπανία είναι, διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, έχουμε διαφορετικέ ανάγκε και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό που η κυρία Μποναφέ ε, προσάρμοσε το κείμενό τη στις ανάγκες μας. Ο κανονισμό αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε αυτή την ευελιξία. Σε κάθε περίπτωση όμω κύριε Βέλα χρειαζόμαστε μια οδηγία για μολυσμένα εδάφη. Ε, η πρόεδρο που θα διακόψει την ομιλήτρια. Το πρόβλημα ξεκινάει στο έδαφο και στο υπέδαφο. Πότε θα έχουμε αυτή την οδηγία, κύριε Βελά. Παρακαλώ πολύ να σέβεστε το χρόνο το οποίο σα ε, δίνουμε. 1,5 λεπτό στον κύριο Χότιμαν εκ μέρου των ε, τον κύριο με εκ μέρους των Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια πολύ σημαντική αυτή η έκθεση, όπως είδαμε πέρσι το καλοκαίρι. Το νερό δεν είναι κάτι το αυτονόητο και πολλέ περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπισαν ξηρασία. Οπότε καταγκάστηκαν να καταφύγουν σε υπόγεια ύδατα για την ε, άρδευση. Λοιπόν, ο κανονισμός αυτός ε, μπορεί να συνεισφέρει πολύ 6,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι στην διάθεσή μας αν μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Βεβαίω ε, πρέπει να έχουμε αυστηρά κριτήρια για να εκμεταλλευτούμε, για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των ε, τροφίμων. Και βεβαίω ε, το θέμα είναι και το τι θα γίνει με τι προτεραιότητε για του αγρότε για να ξαναχρησιμοποιήσουν τα ύδατα. Βεβαίω αυτή τη στιγμή υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν ήδη νερό από τα λίμματα. Τα προϊόντα λοιπόν τα οποία παράγουν οι χώρες ήδη με καθαρισμένο νερό ε, απολύματα καταλήγουν σε χώρες, ε, σε σούπερ μάρκετ χωρών που δεν επιτρέπουν αυτήν την ε, χρήση. Για να προλάβουμε λοιπόν προβλήματα με την στρέβλωση του ανταγωνισμού θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σένρα Ροντρίγκε